ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις διοργανικές πριν από την πρώτη ανάγνωση του Συμβουλίου με βάση το άρθρο 69. Οι θέσεις του Κοινοβουλίου στην πρώτη εντολή αποτελούν ακριβώς την πρώτη ανάγνωση, αποτελούν την πρώτη εντολή και βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ολομέλειας και θα δημοσιευθούν στα επόμενα πρακτικά.